Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία. Αυτό που θα ψηφίσουμε, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που καταφθάνουν και κάθονται. Πού θέλεις να καθίσεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε δύο κείμενα. Πρώτα απ' όλα για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος εποπτείας των συνόρων, ελέγχου των συνόρων. Ο Γιάν Μούλτερ είναι ο εισηγητής. Πριν ξεκινήσουμε η ψηφοφορία, θα ήθελα να σας πω ότι η τροπολογία 174 έχει αποσυρθεί και υπάρχει και ένα, σφάλμα στο κατάλογο ψηφοφορίας όσον αφορά την αιτιολογική σκέψη 7. Τροπολογίες 69 και 67 αναφέρονται σαν ταυτόσιμες αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την 68 και σε περίπτωση που δεν εγκριθεί 68 θα ψηφίσουμε την 69 και μετά την 67. Θα δούμε καθοδόν τι θα γίνει. Θέλει ο εισηγητής να πει κάτι? Όχι. Ο εισηγητής δεν θέλει να πει τίποτα, άρα ας ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Αν είμαστε όλοι έτοιμοι, αν είστε έτοιμοι, να προχωρήσουμε το εγχείρημα της ψηφοφορίας, να Περιμένουμε μέχρι καθίσει συνάδελφος Μπορσελίνο. Οπότε είμαστε σχεδόν όλοι εδώ. Η πρώτη τροπολογία είναι η 49. Ξεκινάμε λοιπόν υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Θα κάνουμε έλεγχο, διεκτονικό έλεγχο. Λοιπόν, Iniziamo con il voto. Voto Πέρας λοιπόν ψηφοφορίας ηλεκτρονικής. Εγκρίνεται. Okay. Εγκρίθηκε λοιπόν η συμβαστική τροπολογία. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές η ίδια ισορροπία ψήφων, αλλά θα κάνουμε επαλήθευση ηλεκτρονική. Πέρασε η συμβαστική λοιπόν τροπολογία. Μάλλον ψηφίσαμε 25-22 ενεκρίθη. 25-22. Εμενταμέντο νούμερο 86. 86. Υπέρ. Κόντρο. Κατά. Αστενούτη. Αποχές εγκρίνεται. 87. 87 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά συμβιβαστική 3 Approvato il compromesso numero Εγκρίνεται λοιπόν η συμβιβαστική 3. Τροπολογία 90 υπέρ. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. με την ίδια ισορροπία εγκρίνεται με τη διαφορά ψήφων. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά αποχές δεν εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ κατά εγκρίνεται. Κομπρομέσο νούμερο Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται η συμβαστική 5. Τροπολογία 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν εγκρίνεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές δεν εγκρίνεται. 105 και προπολογισμών 11 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 106. Υπέρ. Κατά. Δεν εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Προϋπολογισμόν 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 112 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 13 υπέρ κατά αποχές θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Έληξη ψηφοφόρια. Απερίφθη η τροπολογία. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 116 υπέρ 116 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 125. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές δεν εγκρίνεται 17 18 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 133 υπέρ κατά αποχές δεν εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 145. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 150 Πέρας ψηφοφορίας 1831 απερίφθη υπέρ, 151 κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 154 και 155 είναι ταυτόσιμες, ψηφίζουμε μαζί, 154-155 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στη συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται διότι πρόεδρος. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 166. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 167. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 168. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 174 έχει αποσυρθεί. Η τροπολογία 174. Τροπολογία 26 εδώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ κατά απορρίπτεται. 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 και 30 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 183. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 184. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 190. 190. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, λέει ο Θα κάνουμε... Εγκρίνεται. 193 και 194 μαζί ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 196 υπέρ καταπίπτει διότι ενεκρίθη 195 συμφιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 203 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 34 μαζί με τη 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 214 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 218 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 223 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 227, 227 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 228 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 229 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 231 και 232 μαζί υπέρ κατά Αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 235 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.37 έχει αποσυρθεί. 2.36 υπέρ. Σηκώστε τα χέρια παρακαλώ. Κατά. Αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 236. Concluse le operazioni di voto. Πέρας. Rigettato. Περίφ... 238. 238. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται, λέει ο Πρόεδρος. 239. 239. 239. Έντζο. Κύριε Έντσου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 240. Υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 241 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 242 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 243 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 245 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 246 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 247 καταπίπτει. 248 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 249 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 250 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 καταπίπτει 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 253 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ τροπολογία 41 υπέρ κατά από εγκρίνεται Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 259 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Καταπίπτει 260. 261 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στη 44. Πάμε τώρα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 263 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 264 σαν προφορική τροπολογία του εισηγητή. Βλέπετε το κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 265 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 22 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 277 και 278 μαζί. Υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνονται. 279 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 καταπίπτει. 281 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προϋπολογισμών 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμών 4 υπέρ. καταπίπτει, καταπίπτει. Και 4 και 50 καταπίπτει. Και πάμε στην 52 που είναι συμβατή υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 53. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 58 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 του συγκητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 69. Υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Σηκώστε τα χέρια. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 70 υπέρ. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71 και 72 μαζί υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνονται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Προπολογισμών 6 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. προϋπολογισμόν 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. προϋπολογισμόν 8 υπέρ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμόν 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίος 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προϋπολογισμόν 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2 των προϋπολογισμών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προϋπολογισμόν 3. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με το ηλεκτρονικό σύστημα. Il voto si appresta ad essere concluso. Σχεδόν τελειώσαμε, ολοκληρώνει την ψηφοφορία. Καλώς. Πέρας ψηφοφορίας. «51 ψηφίσαντες, 37 υπέρ, 5 κατά, 9 αποχές». Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή. voto. Diamo la parola. La, la, L'onorevole Wikstrom. Συνάδελφε Wikstrom, ζητήσατε να παρέμβετε. Και μετά η συνάδελφος Ματιέ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, μην ξεχνάτε ότι το Σεπτέμβριο είχαμε ψηφίσει ε, για την ουσία, την πολιτική ουσία του κανονισμού του Δουβλίνου και έκτοτε καταβάλουμε άοκνες προσπάθειες να συμφωνήσουμε και για την επιτροπολογία. Βέβαια, τα λόγια είναι πολύ πιο εύκολα από τα έργα, αλλά τελικά αργά το απόγευμα στις 14 Νοεμβρίου καταλήξαμε σε συμφωνία και για την επιτροπολογία. Και μάλιστα η συμφωνία επιβεβαιώθηκε και από τα τρία θεσμικά όργανα. Αυτό που ψηφίζουμε σήμερα είναι το κείμενο που έχουμε συμφωνήσει μαζί με την επιτροπολογία που τελικά εγκρίναμε και ενέκρινε σήμερα και η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσωπιών. Πριν από μία-δύο ώρες εγκρίθηκε και από την Κορεπέρ το θέμα της επιτροπολογία, από τα κράτη-μέλη δηλαδή. Και μετά τη σημερινή ψηφοφορία θα στείλουμε επιστολή, ο πρόεδρο μας θα στείλει επιστολή στο Συμβούλιο, δηλώνοντας ότι αν το Συμβούλιο δεχθεί το κείμενο αυτούσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συστήσει την έγκρισή του χωρίς τροπολογίες στη δεύτερη ανάγνωση. Έμαθα όμως ότι γίνονται κάποιες κινήσεις εντός του Συμβουλίου να παγώσει ο κανονισμός του Δουβλίνου και η οδηγία για τις ε, ε, συνθήκες ε, υποδοχής μέχρι ότου ψηφίσουμε ταυτόχρονα και τα τέσσερα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Δυστυχώς δεν είχαμε ενημερωθεί έγκαιρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις κινήσεις αυτές και σίγουρα δεν έγινε επίσημα κανένα διάβημα. Βέβαια δεν θέλω να στηριχτώ σε εφημολογίες, ούτε να πιστέψω ότι κάποιοι συνάδελφοι θα γίνουν θύματα χειραγώγησης με τέτοιο τρόπο. Οπότε αν έχουμε εκπρόσωπο του Συμβουλίου θα ήθελα να παροτρύνω θερμά την έγκριση του κανονισμού του Δουβλίνου, με το που θα λάβετε την επιστολή μας από τον Πρόεδρο και να μην επιτραπούν άλλες ολιγορίες. Οποιαδήποτε άλλη δράση αποτελεί μια ανέντιμη καταγγελία της συμφωνίας και παραβίασή της. Γιατί χρόνια ολόκληρα ε, διαπραγματευόμαστε το θέμα αυτό. Ήμουν αρχικά πριν από 3,5 χρόνια συγκεντρία και τώρα καταλήξαμε σε ένα κανονισμό που περιλαμβάνει πολύ καλύτερα εχέγγυα για τους ετούντες άσυλο και σαφείς κανόνες για τις ευθύνες μεταξύ των κρατών μελών. Είναι σημαντικό να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός άνευ χρονοτριβής. Γι' αυτό και ζητώ σας παρακαλώ για την υποστήριξή σας. Και μην ξεχνάτε και τη προθεσμία του 2012 θα είναι αδύνατον να τηρήσουμε την προθεσμία αυτή αν δεν εγκρίνουμε σήμερα και το Συμβούλιο δεν εγκρίνει τον κανονισμό. Γιατί έχουμε πολλούς ευάλωτους ανθρώπους που πατάνε το ευρωπαϊκό έδαφος. Δεν θα πρέπει να μελούμε την κατάστασή τους. Η κυρία Ματιέ. Διαπιστώνω ότι όλοι ε, βιαζόμαστε να ψηφίσουμε. Το ίδιο και το ΕΛΚ και εμείς ε, θέλουμε να ψηφίσουμε το συντομότερο δυνατόν και γι' αυτό είπαμε να ψηφιστεί ως τμήμα του πακέτου και η Eurodac και μάλιστα ζητήσαμε σήμερα ψηφοφορία για την ε, έκθεση παρόλο που διαφώνησαν οι υπόλοιπε πολιτικές ομάδες και δεν ε, δέχτηκαν να ψηφίσουμε νωρίτερα για την ε, Eurodac 17 Δεκεμβρίου. Θεωρούμε ότι και η Eurodac αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα του συνολικού πακέτου και είναι λογικό να ψηφιστούν από κοινού αυτά τα θέματα. Είχαμε ζητήσει να ψηφίσουμε για την Eurodac 17 και 18 Δεκεμβρίου. Απορρίφθηκε το έτοιμά μας, γι' αυτό και τελικά αποφασίσαμε να απόσχουμε στην ψηφοφορία που θα ακολουθήσει. Καλώς. Υπενθυμίζω σε όλους σας ότι θα ψηφίσουμε είναι θέλουμε να δούμε τα κριτήρια και μηχανισμούς του καθορισμού του αρμοδίου κράτους μέλους για την εξέταση ενός αιτήματο διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα από τα κάτι μέλη από έναν πολίτη ε, τρίτης χώρας ή από έναν Ε, λοιπόν, μπορούμε να ψηφίσουμε. Υπέρ. ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λοιπόν, πέραση ψηφοφορία. Non Αντιπρόεδρος δεν ψηφίσατε. Η γραμματεία σημειώσει και να καταχωρηθεί ψήφος. 18 υπέρ, 5 εκατά, 25 αποχές. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Μπορούμε να κάνουμε την υπόλοιπη δουλειά. Το δικαίωμα της πρόσβασης είναι το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Όποιος δεν ενδιαφέρεται, πώς να το πω, μπορεί να ακολουθήσει άλλη κατεύθυνση. Μιλάμε λοιπόν για το δικαίωμα πρόσβασης σε υπεράσπιση όσον αφορά τα ποινικά ζητήματα δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. και δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη. Η συγγήτρια είναι η κυρία Έλενα Οάνα Αντωνέσκου. Προστασία λοιπόν και προστασία των, πάντα των διαφόρων ε, δικαιωμάτων αυτών, πάντα αυτό το θέμα. Παρακαλώ, αν θέλετε να μιλήσετε κάποιοι, παρακαλώ να βγείτε από την αίθουσα. Λοιπόν, πάντα ήταν ε, βασικό, βασική μέρημνα τη ε, πολιτική του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Το είδαμε και στι διαπραγματεύσει που κάναμε για την οδηγία για την ερμηνεία στις ποινικέ διαδικασίες και την ενημέρωση στις ποινικέ διαδικασίες. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών εργάστηκε άκναμπη του θέματος και ήθελε να υπάρχει το ύψιστο επίπεδο προστασίας όσον αφορά τα μέσα που θετούνται. Γίνονται τώρα τα διαπραγματεύσει ε, διαδικασία αυτή που αφορά το δικαίωμα πρόσβαση δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και δικαίωμα επικοινωνία μετά τη σύλληψη διαπραγματεύσεις ε, γίνονται στο Συμβούλιο που εκπροσωπείται από την Κυπριακή Προεδρία. Τρεις τριμερείς διάλογοι έγιναν, ο επόμενος προβλέπεται να διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου του έτους αυτού. Ε, Στρέφουμε προς την κυρία Αντωνέσκου, ούτω ώστε να μπορέσει να μας παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί στον φάτη της διαπραγματεύσεις και τα επιτευθέντα αποτελέσματα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πρώτα από όλους συναδέλφους την πρόταση οδηγίας ε, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που έχει ως ε, αντικείμενο την αποκατάσταση των δικαιωμάτων ε, για ε, κατηγορούμενους σε ποινικέ δίκη Το δικαίωμα επικοινωνία, το δικαίωμα πρόσβαση ε, σε δικηγόρο, το δικαίωμα επικοινωνίας με έναν τρίτο, είτε είναι μέλο αυτό τη οικογένεια, είτε όχι. Η πρόταση αυτή συνιστά ένα επιπλέον βήμα μετά το ψήφισμα το 2009 σε σχέση με τα δικονομικά δικαιώματα των ε, κατηγορουμένων. Ενδέστε στο πρόγραμμα της Στοχόλμης που ενέκρινε το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2010. Και όπως ε, έχει δηλώσει το Συμβούλιο, στις 8 Ιουνίου υιοθετήθηκε μία ε, θέση για το θέμα αυτό μετά την υποβολή της πρώτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από ε, μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις έχουμε μια κατάληξη. Βέβαια οι χρονοβόρες διαπραγματεύσεις δικαιολογούνται από την ευαισθησία αυτού του θέματος σε ένα θέμα ε, για το οποίο υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών. Δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση για το πώς θα πρέπει να ερμηνευθεί και η ευρωπαϊκή νομολογία. Και στην ε, ψηφοφορία προς ανατολισμού που είχαμε τον Ιούλιο στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ε, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις που ε, ξεκίνησαν τον ε, Σεπτέμβριο. Είχαμε τρεις τριμερείς διαλόγους και συναντήσεις με τους ασκιώδεις συγητές και τεχνικές συζητήσεις. Στους τρεις τριμερείς διαλόγους εξετάσαμε τα 7 πρώτα άθρα της πρώτης οδηγίας και είχαμε και συζητήσεις για το πεδίο εφαρμογής, για το στόχο, το δικαίωμα ε, εκπροσώπηση από δικηγόρο, το δικαίωμα επικοινωνίας μετά την σύλληψη, το δικαίωμα επικοινωνίας με προξενικές ή διπλωματικές αρχές γενικώ και το δικαίωμα για τα απόρριτα, δικαίωμα απόρριτα δεδομένα, απόρριτα στοιχεία. Συνεχίζονται βέβαια οι συζητήσεις και θα συνεχιστούν και στο μέλλον γιατί έχουμε μείνει κάποιες εκκρεμότητες ε, για ορισμένα άρθρα. Θα συνεχιστούν λοιπόν οι διαπραγματεύσεις και στη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας και οι συζητήσεις ε, δεν θα σταματήσουν. Τώρα υπάρχει ένα άρθρο, ένα άρθρο που αφορά του ε, τους ε, που δεν είναι υποπτοί για παράδειγμα το δικαίωμα ε, για ένδικη προστασία, για άσκηση προσφυγής, για διατήρηση επίπεδου προστασίας, αλλά και ε, ένα άρθρο που αφορά την εσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κυπριακή Προεδρία για τις άοκνες προσπάθειές της ε, στον τομέα αυτό κατά τη διάρκεια των τρίμηνων διαπραγματεύσεων. Είχαμε, όπως σας είπα, πολλές τεχνικές ε, συναντήσεις ε, και επαφές με τα κράτη-μέλη. Υπάρχει αισθητή πρόοδος, ε, διαπιστώνεται από τους ενδιαφερομένους και το κείμενο σε μεγάλο βαθμό διαφέρει πια αρκετά από το κείμενο που είχε εξεταστεί και ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μας ε, βοηθάει με τις δικές προσπάθειες και την υποστήριξή της. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω αλλά να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και για τις προσπάθειες που κάναμε όλοι από κοινού. Επαναλαμβάνω, πολύ άριθμες ήταν οι συναντήσεις και οι συνεδριάσεις και ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα συνεχιστεί αυτή η αξιοθαύμαστη συνεργασία. Μέσα σε ένα τρίμηνο σημειώσαμε αρκετή πρόοδο, αλλά θα χρειαστούν και περαιτέρω συζητήσεις για να καταλήξουμε στη συμβαστική λύση. Προσωπικά πάντως πιστεύω ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα ήθελα να καθησυχάσω τους συναδέλφους διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν θα αφήσω προσπαθειών προκειμένου αυτό το σημαντικό νομοθετικό εργαλείο για τα δικονομικά δικαιώματα των κατηγορουμένων να ε, τελεσφορήσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα ε, και έντονος ο ρυθμός των εργασιών, αλλά ευελπιστώ ότι με τη συνεργασία όλων θα καταλήξουμε σε αίσια αποτελέσματα. Ευχαριστώ, Άννα. Να δώσω το λόγο μετά από αυτή την παρουσίαση τη λεπτομέρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Κνούτσεν και ο κύριος Ολιβερτέλ ή κάποιος άλλος που αντιπροσωπεύουν αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ε, thank you very Ευχαριστώ πολύ. Υπογραμμίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συμβιβαστική λύση πάνω σε μια οδηγία ισορροπημένη και αποτελεσματική για τα δικαιώματα πρόσβασης σε δικηγόρο ε, και επικοινωνίας. Ε, επετελέστη πρόοδος κατά τον τριμερή διάλογο μέχρι τώρα και προσωπικά ευχαριστώ την κυρία Αντωνέσκου και την ομάδα της για τις πολύ σημαντικές προσπάθειες ε, που έκανε. Και πράγματι οικοδομήσαμε καλές σχέσεις εργασίας με όλα τα μέρη. Ελπίζουμε ότι αυτή η δυναμική θα μπορέσει να διατηρηθεί στις συζητήσεις για αυτό το σημαντικό φάκελο, ελπίζοντας ε, ε, ότι με τον σωστό προβληματισμό και δέσμευση όλων των μερών θα συμφωνήσουμε σε ένα κείμενο υψηλής ποιότητας και προτύπων ε, προστασίας στο άμεσο μέλλον, στο, μισό, στο πρώτο μισό της Ιρλανδικής Προεδρίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνεχίσει να υπολογίζει στην ισχυρή δέσμευση της Κομισιόν που θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την εισηγήτρια και με τους κοιόδης επίσης για την επίτευξη της συμφωνίας αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν η Κυπριακή Προεδρία δεν είναι, δεν έχει εκπρόσωπο. Μπορούμε να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους που ζήτησαν. Κύριος Κίρκοπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ καταρχήν ε, την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά. Δεν, ε, δεν μιλώ μόνο ως βουλευτής αλλά και ως δικηγόρος και πράγματι συζήτησα το μέτρο αυτό με τον πρόεδρο της ε, Νομικής Ένωσης στο Λονδίνο πριν από λίγες μόνο ημέρες και θέλω να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Σημαντικές κινήσεις του πληθυσμού με τα ταξίδια στην Ευρώπη ε, επηρεάζουν τη σημασία του θέματος. Βέβαια γιατί θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος δικηγόρος ε, πάντοτε. Αλλά πάντοτε ε, οι Βρετανοί πολίτες που πηγαίνουν στην Ισπανία για παράδειγμα είναι 13 εκατομμύρια και 2.000 από αυτούς ε, δυστυχώς θα συλληφθούν διότι διέπραξαν, είναι ύποπτοι ότι διέπραξαν αξιόπινη πράξη. Δεν είναι κάτι που μας κάνει περήφανος αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό στα δικαιικά συστήματα που αναμφισβήτητα έχουν διαφορές οι άνθρωποι να έχουν σωστή εκπροσώπηση το ταχύτερο δυνατόν από έναν επαγγελματία που γνωρίζει το σύστημα και μπορεί να τους παράσχει αρρωγή στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Γιατί δεν είναι οι 2.000 ένοχοι για κάτι, χρειάζονται βοήθεια όμως. Και άλλες χώρες ε, έχουν παρόμοιο, παρόμοιο σύστημα. Είναι δύσκολο το θέμα γιατί δεν έχουμε κοινό ποινικό σύστημα. Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες. Πόσο, ε, πόσο μάλλον είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει εκπροσώπηση από δικηγόρο. Επίσης ε, θα πρέπει να γίνει σεβαστή εμπιστευτικότητα. Δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα καθ' αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό στην επικοινωνία μεταξύ κάποιου που είναι ύποπτος και του δικηγόρου του, όσο είναι δυνατόν οι συζητήσεις θα πρέπει να είναι φύσεως εμπιστευτικής. Ε, Εμεί επίση θέλουμε να υπάρχει πρόσβαση και από το τηλέφωνο, αν δεν μπορούν να είναι εκεί παρόντε, να έχουν φυσική παρουσία οι δικηγόροι. Καλύτερο από το τίποτα. Και το θέμα του κόστου, η νομική ε, αρρωγή ε, δωρεάν έχει επίσης ε, τύχη χωριστής επεξεργασίας, αλλά και αυτό θα στοιχίσει 32 ή 33 εκατομμύρια στερλίνες για να εφαρμοστεί. Δεν είναι σημαντικό το ποσό, γιατί βέβαια αυτή τη στιγμή όλοι για τον προϋπολογισμό μιλάμε. Δεν είναι μεγάλο το ποσό λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη υποστήριξη που μπορεί να παράσχει το σύστημα και τέλος, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι όλοι μας πολύ σωστά ανησυχούμε να μην αφήσουμε απομονωμένους τους πολίτες μας σε καταστάσεις που δεν μπορούν να φροντίσουν για τα δικαιώματά τους. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα η εκπροσώπηση και η υποστήριξη. Ε, εν πολλής είμαστε υπέρ Πιστεύουμε ότι ήταν αξιέπαινο το έργο της εισηγήτριας και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η δική του στάση ε, είναι υποστηρικτική, άρα και αξιέπαινη επίσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Κυρκόπ. Συνάδελφε Άλμπρεχτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, συμφωνώ μετά όσα είπε ο κύριος Κέρκοπ λαμπρό το έργο του, της συγγήτριας. Μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Η συγγήτρια εργάστηκε πολύ σκληρά και εργάζεται για να πετύχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και ευχαριστώ πολύ για την ε, πολύ καλή συνεργασία με τους κοιόδης συγγητές. Είμαστε σε καλή πορεία. Μου αρέσει η πρόοδος που έχουμε πετύχει και το πώς προχωράμε. Ξεκινώντας από όσα είπαν οι προλαλήσαντες, μπορώ να πω ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα αν δεν δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι πολύ δυσνόητο και περίπλοκο. Είναι ένα απλό δικαίωμα, εύληπτο το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, πρόσβασης σε δικηγόρο, σε όλες τις όταν, κάποιο, όταν είμαι ύποπτος, όταν μου απαγγέλλεται κατηγορία. Έπρεπε να είναι κάτι απλό, να μην περιέχει πολλές παρεκκλήσεις και εξαιρέσεις. Πάνω σε αυτή τη βάση πρέπει να κινούμεθα. Να μην προσπαθούμε να λύνουμε πάντα, να καλύπτουμε όλες τις τυχόν ερμηνείες που θα μπορούν να δώσουν οι δικαστές κατά κάθε υπόθεση. Να μην επιλύουμε κάθε περίπτωση στην νομοθεσία. Δεν είναι σωστή προσέγγιση. Και γι' αυτό ζητώ από το Συμβούλιο και από κάποια κράτη-μέλη που θέλουν να δουν, να αντικατοπτρίζεται το δικό τους νομικό πλαίσιο στην οδηγία, να είναι πιο ανοιχτά. Να υπάρξει αυτό το κοινό νομικό πλαίσιο που δημιουργείται από αυτή την οδηγία, με έναν στόχο τελικά, την εφαρμογή της αρχής της δίκαιης δίκης που έχουμε στο άρθρο 6 της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα να υλοποιείτε, να ακολουθείτε αυτό και στην Ομοθεσία των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Πρέπει αυτό να το καλύπτουμε και να το επιτυγχάνουμε μέσω της οδηγίας και ζητώ από τα κράτη-μέλη κυρίως όσον αφορά τον εμπιστευτικό χαρακτήρα ε, της συνομιλίας του υπόπτου με το δικηγόρο. Αυτό να εξασφαλίζεται. Είναι σημαντικό κομμάτι. Να μην υπάρχουν εξαιρέσεις για μικρά παραπτώματα που ίσως δημιουργούν αμφιβολίες και προβλήματα. Τι σημαίνει αυτό το μικροπαράπτωμα, το μικροαδίκημα. Μπορεί να ακολουθείτε σοβαρή διαδικασία, να μην μπλέκω σε μια διαδικασία ποινικού δικαίου χωρίς δικηγόρο. Και θα πρέπει να ταιριάζει και η προσέγγιση με την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. να μην γίνεται επικοινωνία με το δικηγόρο μέσω ε, αλληλογραφίας και μέσω τηλεφώνου. Υπάρχει πραγματική παρουσία του δικηγόρου εκεί. Να συμμετέχει στη διαδικασία, να μην παρακολουθεί από μακριά τι συμβαίνει, να μπορεί να δρά, να κινείται υπέρ του πελάτου του ο Αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό στο νομικό πλαίσιο που φτιάχνουμε και παρεκκλήσει, εξαιρέσει. Όταν χρειάζεται κατά περίπτωση απόφαση ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόσβαση για δικηγόρο, αυτέ οι εξαιρεσει να είναι πολύ περιορισμένες, πολύ λίγες. Πρέπει να επιμείνουμε έναντι του Συμβουλίου πάνω σε αυτά και έχουμε τα κατάλληλα επιχειρήματα. Μιλάμε για ελάχιστες απαιτήσεις αυτές, πραγματικά ελάχιστες. Και τα κράτη-μέλη μπορούν να προχωρήσουν πιο πέρα. Αυτό ζητά λοιπόν, μας ζητείτε να εφαρμόσουμε και θα πρέπει να επιμείνουμε όταν θέλουμε να συμμορφωθεί λοιπόν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Βούς. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόσβαση στο σύστημα δικαιοσύνης είναι πολύ σημαντικό, το είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι ούτω ώστε να αντιμετωπίζονται δίκαια οι άνθρωποι που θεωρούνται ύποπτοι ή διέπραξαν μια αξιόπινη πράξη σύμφωνα με το, τις συνταγματικές επιταγές κάθε χώρας. Θα πρέπει να εντάσσεται στη διαδικασία από, την αρχή ο δικηγόρος. Γι' αυτό ε, προτείνει η συγγήτρια φιλόδοξες λύσεις, σωστές λύσεις και χαίρομαι που η συγγήτριά μας Ιωάννα τα επεξεργάστηκε αυτά πολύ λεπτομερώς και ασχολήθηκε με, όλα, με όλες αυτές τις λεπτομέρειες και προσπαθεί τώρα να περάσει τις προτάσεις της διαπραγματεύσεις. Εγώ θέλω μόνο να ρωτήσω αν σε αυτά τα σημεία ε, υπάρχουν προϋποθέσεις ευθύνης και θέμα εμπιστευτικότητας και αν στις διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει τα θέματα αυτά, ούτως ώστε να διαφαίνεται προς τα που πηγαίνει η κατεύθυνση της συζήτησης. Η ε, κυρία Ματιέ, ευχαριστώ. Καταρχήν συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας, γιατί επέδειξε ύψιστη επαγγελματική συνείδηση και μεγάλη αποτελεσματικότητα και η πρόοδος που σημειώσαμε οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις δικές της προσπάθειες. Την ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις ως προς εξαιρέσεις που ανέφερε η συγγήτρια. Η δική μου ανησυχία που την παρουσίασα και στην Συγκεντρική και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά τις εξαιρέσεις και ιδιαίτερα για όσους έχουν κατηγορηθεί για τρομοκρατικές πράξεις. Ε, συμφωνώ με την πρόταση του κυρίου Άλμπερχτ σε ό,τι αφορά τι για τα πτέσματα ή τα μικρά παραπτώματα, αλλά για τις σοβαρέ περιπτώσεις ε, αποδεδειγμένης τρομοκρατική ενέργειας θα μπορούσα, καλό θα ήταν να επιτρέπονται εξαιρέσεις για την ταχύτητα της έρευνας και για να μην παραβλάψουμε την ποιότητα του έργου της αστυνομίας σε περίπτωση τρομοκρατικών ενεργειών και βίων θανάτων. Ε, θα ήθελα λοιπόν η συγκεκριά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πούν τι γίνεται με το συγκεκριμένο σημείο. Επίσης θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις από την εισηγήτρια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το χρονοδιάγραμμα. Μπορούμε έστω και κατά προσέγγιση να έχουμε ενδείξεις για το χρονοδιάγραμμα γιατί είναι πολύ σημαντική έκθεση. Και τι γίνεται με την δικαστική αρρωγή, θα μπορούσε να μας πει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί το είχαμε αναφέρει αυτό. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι η κυρία Ρέντινγκ δεν ήθελε να συνδέσει τις δύο προτάσεις, να υποβάλει την πρόταση για το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο και τις, το θέμα της δικαστικής αρρωγής, αλλά θα ήθελα να δω πώς προχωρούν τα πράγματα, να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προχωρούν τα πράγματα σε αυτό το θέμα. Η κυρία Ρομέρα Λόπες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, Πρόεδρε, σε αυτή την πρόταση οδηγίας να τονίσω το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο αναφέρεται στι περιπτώσει που ο ύποπτο ή κατηγορούμενος μπορεί να αναλάβει το κόστος, γιατί δεν μιλούμε για δωρεάν δικαστική, ε, παρουσία δικηγόρου. Και στο μέτρο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σημειώσει κάποια πρόοδο για μια δωρεάν τέτοια δικαστική αρρωγή, για παρουσία δωρεάν, δωρεάν παρουσία δικηγόρου, τότε το δικαίωμα αυτό θα έχει πολύ περιορισμένη εφαρμογή. Μια και θα πρέπει να μπορεί να αναλάβει τα δικαστικά έξοδα ο κατηγορούμενο ή ύποπτο. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τέτοια πρωτοβουλία να αναλάβει για να υλοποιηθεί αυτό το δικαίωμα πρόσβαση σε θα πρέπει να είναι δωρεάν αυτή η συνδρομή. Γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Ε, σε μερικές χώρες η δωρεάν ε, ε, συνδρομή δικηγόρου είναι πολύ περιορισμένη και έτσι δημιουργούμε διαφορές μεταξύ πλούσιων και φτωχών κατηγορουμένων ή υπόπτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το οδικό χάρτη για τις ε, δικαστικέ ε, εγγύησεις έχουμε δύο δικαιώματα. Το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο και το ε, δικαίωμα επικοινωνία στη στιγμή της κράτησης. Αρχικά ήταν ανεξάρτητες αυτές οι δύο εγγύησεις. Θα ήθελα να εξάρω τι τεράστιε προσπάθειες τη εισηγητρίας και να τι συγχαρώ για αυτές, γιατί αφαιρέσαμε τα λιγότερα προβληματικά θέματα και προχωρήσαμε σε πολλά από αυτά. παράδειγμα, την προέλευση του δικαιώματος και τη στιγμή γέννησης του δικαιώματος. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και χάρη στην εισηγήτρια προχωρήσαμε, αλλά εκκρεμούν πιο επίμαχα ζητήματα. Το θέμα των εξαιρέσεων, για παράδειγμα. Η χώρα μου έχει μία μακροχρόνια παράδοση αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και πολλές φορές ε, γίνονται κάποιες καταχρήσεις ε, με άλθη την αντιτρομοκρατική πολιτική και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη δεν μόνο το θέμα των εξαιρέσεων, αλλά και το θέμα της παρουσίας του δικηγόρου σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων και το ρόλο του δικηγόρου. Επίσης, το δικαίωμα, η εμβέλεια τη, των δραστηριοτήτων του δικηγόρου για να εξασφαλιστεί πραγματικά αποτελεσματικό δικαίωμα υπεράσπιση. επίση περίοδο επικοινωνία και το δικαίωμα σε δικηγόρο, ακόμη και αν δεν είναι η πρώτη επιλογή του ενδιαφερόμενου και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά αυτά είναι πιο ευαίσθητα ζητήματα το θέμα, το, το θέμα των πτεσμάτων ή των λιγότερο σοβαρών ε, αδικημάτων. Θα ανακύψουν αυτά αναγκαστικά στην πορεία. Επειδή το θέμα είναι δύσκολο, προτιμώ να μην βιαστούμε, γιατί καλύτερα να έχουμε μια καλή οδηγία παρά να τορπιλήσουμε τη συμφωνία εξαιτία υπερβολική σπουδή. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα των δικονομικών εγγύσεων και αυτό καλύτερα να βαδίσουμε αργά αλλά σταθερά. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσίπελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα, θέλω να μιλήσω πάνω σε δύο θέματα. Πρώτον, πάντοτε με συγκλονίζει όταν μαθαίνω σε ποιους τομείς χωρίς ε, να κουνήσουμε το βλέφαρο, δίνουμε εκατομμύρια, ε, ενώ όταν πρόκειται για σημαντικά θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, μας απασχολεί ξαφνικά το κόστος, σκεφτόμαστε την κρίση και λέμε ότι δεν επιτρέπεται να δαπανίσουμε τα χρήματα αυτά. Ε, δεν ανταποκρινόμαστε έτσι στη θεμελιώδη σημασία του θέματος. Τέλος, για τις εξαιρέσεις, στο δεύτερό μου θέμα. Πρόκειται εδώ για σημαντικά θεμελιώδη δικαιώματα και ανθρώπους των οποίων η ενοχή πρέπει να ε, αποδειχθεί γιατί όποιος προσάγεται στο δικαστήριο δεν είναι ένοχος. Το να αρχίσουμε με τις εξαιρέσεις θεωρώ ότι είναι ανεύθυνο και δεν ισχύει μόνο για μέσης σοβαρότητος αδικήματα αλλά και για την τρομοκρατία. Ξέρουμε από όλες συζητήσεις στο παρελθόν ότι δεν είναι όλοι ένοχοι όσοι κατηγορούνται για τρομοκρατικές ενέργειες, ούτε καταδικάζονται όλοι. Καμιά φορά στο τέλος της διαδικασίας διαπιστώνεται μάλιστα η αθωότητά τους. Ιδιαίτερα σε μια τέτοια σοβαρή περίπτωση να στερήσουμε το δικαίωμα στον ύποπτο, το δικαίωμα να έχει ένα δικηγόρο, θεωρώ ότι είναι εντελώς ανεύθυνο. Νομίζω ότι ο κύκλος των παρεμβάσεων από πλευρά συναδέλφων εξαντλήθηκε επανειλημμένα αναφέρθηκε η συνάδελφος Αντωνέσκου οπότε της δίνω το λόγο για να ολοκληρώσει τον κύκλο αυτό Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους για την συνεργασία τους και για αυτά που είπαν είδα σε ποιο βαθμό αυτό το θέμα είναι σημαντικό για την Επιτροπή μας και σε ποιο βαθμό οι θέσει των συναδέλφων είναι σωστές και σταθερές, κυρίως όσον αφορά διάφορες συγκεκριμένες στοιχείες της οδηγίας και για μας είναι ένας καλός δείκτης, δείχνει τη δυσκολία που έχει αυτό το θέμα. Όσον αφορά το, την εμπιστευτικότητα των συνομιλιών, Πάντα το θέμα της εμπιστευτικότητας ήταν σημαντικό για το Κοινοβούλιο. Πάντα θεωρούσαμε ότι χρειάζεται η εμπιστευτικότητα. Και στην τελική θέση του Κοινοβουλίου, μετά την αρχή ψηφοφορία, την ενδεικτική, αναφέρθηκε ότι οι συζητήσεις μεταξύ του νομικού και του πελάτου πρέπει να είναι ε, εμπιστευτικού χαρακτήρα. Αλλά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν έχουμε επιληφθεί αυτού του σημείου ακόμα. Το συζητάμε, δεν το ολοκληρώσαμε. Όσον αφορά τις εξαιρέσεις, ε, στη θέση του Συμβουλίου είδαμε ότι προτιμά το Συμβούλιο μια προσέγγιση ε, κατά περίπτωση. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο θεωρεί ότι σε κάποιες συγκεκριμένες περιστάσεις οι εξαιρέσει θα πρέπει να προσαρμόζονται ε, αναλόγως με την κάθε περίσταση. Ε, όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβαση στο δικηγόρο, είναι περιορισμένες οι εξαιρέσει. Όσον αφορά το δικαίωμα της επικοινωνίας, εκεί υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια λιγμών. Σας μιλώ τώρα για τη θέση του Συμβουλίου και όχι για το κείμενο του Κοινοβουλίου. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι συζητήσεις πρέπει να συνεχιστούν όσον αφορά τις εξαιρεσει και θα σας κοινοποιήσουμε το τελικό αποτέλεσμα προφανώς. Αν επιτρέπετε θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτή τη νομική βοήθεια κατά την άποψή μας είναι απαραίτητο να μας πούν οι συνάδελφοι της ε, Κομισιόν σε ποιο στάδιο έχουν φτάσει οι συζητήσεις ε, όσον αφορά τα όσα ζήτησε το, τα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Διότι αυτή η οδηγία ε, δεν μπορεί να διαχωριστεί από το θέμα της νομικής αρρωγής, της βοήθειας. Θα ήθελα λοιπόν να πω τελικά ότι Πρόκειται περί θέματος περίπλοκου. Ε, οι συζητήσεις συνεχίζονται. Ελπίζουμε το τελικό αποτέλεσμα να είναι θετικό και ενθαρρύνω τους συναδέλφους να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους όπως έκανα μέχρι τώρα διότι είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε να πετύχουμε το βέλτιστο δυνατό τελικό αποτέλεσμα. Καλώς, αναμφισβήτητα το σημείο ισορροπίας είναι να πετύχουμε να συσχετίσουμε τα συμφέροντα του, α, του ατόμου που είναι του υπόπτου με τις ανάγκες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει τα διάφορα φαινόμενα, τα εγκληματικά κλπ. Λοιπόν, εμπιστευόμαστε εισηγήτη ότι θα βρει τη σωστή ισορροπία. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας, υπενθυμίζοντας ότι οι επόμενες συνεδριάσεις θα είναι στις 10, στις 10 Δεκεμβρίου. Ε, στο, Στρασβούργο και 17 και 18 Δεκεμβρίου στις ε, Βρυξέλλες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την διερμηνία και την ε, γραμματεία.